τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας, δεν βλέπω αντιρρήσεις και ως εκ τούτου εγκρίνω.